Um, uh, Καλησπέρα σας, λέει ο Πρόεδρος. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίασή μας, που είναι πάρα πολύ μεγάλης ε, σημασίας ε, για το έργο της Επιτροπής. Το πρώτο μας σημείο στην ημέρηση διάταξη είναι η έγκριση της τη διάταξης. Εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, θεωρώ ότι εγκρίνεται και Δεύτερο σημείο, οι ανακοινώσει του Πρόεδρου, οι αποφάσει των εισηγητών τη 24η Σεπτεμβρίου. Κάντε λίγη ησυχία, παρακαλώ. Οι αποφάσεις υπάρχουν στον φάκελο μεταγραφά της συνεδριάσεως, αν δεν έχετε ενστάσεις και ε, αυτές οι αποφάσεις εγκρίνονται. Τρίτο σημείο, Brexit η σχετική συζήτηση της προηγουμένης ε, εβδομάδας, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στην Επιτροπή μας την ε, πρόταση για ε, κανονισμό του Συμβουλίου σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2020. Έτσι θα τον το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και οι δικαιούχοι να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα συνεργασίας εάν και εφόσον συνεχίσει να συμβάλλει στον προπολισμό η χώρα και αν αποδεχθεί τους σχετικούς οικονομικούς και άλλους ελέγχους ε, είναι προς το συμφέρον όλων να εξασφαλιστεί ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα γίνει έφτακτα και κατόπιν συμφωνίας και αυτό το κατεπήγον ε, μέτρο πρόκειται να μας επιτρέψει ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρξει ε, συμφωνία να έχουμε κάποια ε, κανονική ροή των πραγμάτων και γι' αυτό ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εγκρίνει αυτή την πρόταση. Και τώρα δώσω το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, εάν θέλουν το λόγο. Ιδάλλως σε άλλους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν από αυτού. Εάν θέλει κανείς το λόγο, ε, κλείνω λέγοντα ότι τροπολογίε μου υποβληθούν μέχρι τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο σημειώστε ότι η τροπολογία μπορεί να αφορά την πρόταση να απορρίψουμε την πρόταση και από πλευρά τη διαδικασία. Θα γίνει η ψηφοφορία μόνο άπαξ και έχει γίνει η επίσημη παραπομπή του σχεδίου του κανονισμού. Ε, έχει διαβαστεί σε εμάς. Οπότε, ε, από ό,τι γνωρίζω αυτό θα γίνει σύντομα και θα ψηφίσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, ψηφοφορίε. Πρώτα-πρώτα. Να κάνουμε μια δοκιμή. Ψηφίζουμε τώρα. Παρακαλώ πιέστε κάποιο από τα κουμπιά. Της... votes. 34 ψήφισαν ε, πέρα Πάμε τώρα στο σημείο 4 της διατάξεως. List uh, DEP 4. Uh, ε, I give the word to the rapporteur. Σχέδιο προϋπολογισμού. Δώσω το λόγο στον τον κύριο Χάουαρντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να πω το εξής. Να εξηγήσω ότι Έχει αποσυρθεί η τροπολογία 1725 και έτσι υπάρχει κάποια συνοχή περισσότερη στην πρόταση όσον αφορά το ότι θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκε των δεσμικών οργάνων σε περίπτωση αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 31 Οκτωβρίου. Σε αντίθεση με το πρώτο σχέδιο του προπολογισμού που είχε ως βάση την 29η Μαρτίου. Uh, with the vote by uh, hand raising uh, για να δούμε τώρα, ο πρόεδρος. 12, 16. Οι τροπολογίες ποιοι είναι περ, ποιοι είναι κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες στο σχέδιο ψηφίσματος. Amendments Τροπολογίες Υπάρχει προφορική τροπολογία, λέει κάποιος κύριος. Α, αυτό, αυτό εννοούσα. Πρώτη τροπολογία, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται δεύτερη τροπολογία, παραθμόν 2. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 3. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία πέντε Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. έξι Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατονομαστική ψηφοφορία όσον αφορά την τελική έκθεση. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 30 υπέρ και 5 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Χάουαρτ. Πέντε. Ενεργοποίηση του μέσου Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Συγγνώμη, κάνα λάθος λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. άποχέ, Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. άποχέ. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική ε, παράγραφος Δέλτα, πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 30 υπέρ, 4 κατά, με 3 αποχέ εγκρίνεται. 6. Τη ημερία διατάξεω. Μεταφορά πιστώσεων δεν έχουμε και πότε πάμε στο 7. Άλλα θέματα μεταφοράς ε, κονδυλίων και πιστώσεων. Κύριε Φερναντές, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Α, να σας τα πω στα πορτογαλικά. Έχω μια μεταφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλα τμήματα για να ενισχυθεί ε, το ποσό για το 2022. 340.000 ευρώ. Δαπάνες συντήρησης ε, κτιρίων στις Βρυξέλλες. Αυτές οι δαπάνες θα καλυφθούν από την μεταφορά υπολείπου από άλλα, άλλες γραμμές του προπολογισμού. Προτείνω να ψηφίσουμε υπέρ. Thank you. Any of the shadow reporters wants to take the floor. ηγητές θέλουν το λόγο. Όχι. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 6 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Πολιτική κτηρίων, σημείο 8. Κτηριακή πολιτική, δεν υπάρχει κάτι στην ημερήσια διάταξη για αυτό το θέμα, οπότε θα περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 9. Το βασικό θέμα μας για σήμερα Η συνεδρίαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί θα ψηφίσουμε ακριβώς αυτό το κείμενο. Είναι 1.365 τροπολογίες. Στον προϋπολογισμό του 2020 έχουν υποβληθεί από ομάδες, επιτροπές και από μέλη. Κυρία Χολμάγερ είναι η εισηγήτρια και η κυρία ε, Γκαρδιαθάβαλ Ρουβιάλ για τα συνεισηγήτρια. Πάρα πολλέ ώρες και μέρες και μήνε δουλειά κρύβονται πίσω από αυτές τις τροπολογίες, από αυτό το κείμενο. Ειδικά τι τελευταίες εβδομάδε χρειάστηκε να αναλύσουμε και τις συμβιβαστικέ προτάσεις. Θα δώσω το λόγο στι εισηγήτριε για να μας παρουσιάσουν την προσέγγιση τους και τις συμβαστικές προτάσεις. Κύριε Χολμάιερ. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα προσπαθήσω βέβαια να αναλύσω όλες τις 1365 ε, τροπολογίες και τις συνέπειες που αυτές έχουν. Ε, αυτό έχει συζητηθεί και με τους κοιόδης ηγητές, ε, με τη γραμματεία, με όλους τους βοηθούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους όσους μας βοήθησαν. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά και θεωρώ πως καταλήξαμε σε έναν καλό συμβιβασμό. Βέβαια το Συμβούλιο έκανε τα σχέδιά του στην αντίθετη κατεύθυνση από τη δική μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να συμπλέξουμε Ε, πρώτον, περιβάλλον, καινοτομία, life scene και αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτή είναι το οι οποίοι μας απασχόλησαν. Είναι μία ομάδα, μετά υπάρχει και άλλη ομάδα για, ε, τροπολογιών για τους νέους. Έπειτα, αναπτυξιακή βοήθεια, όργανα γειτονίας. Σε αυτούς τους τομείς ζητάμε ενισχυμένους πόρους σε σχέση με αυτά που αποφάσισε το Συμβούλιο. Επίσης, ε, Διαφωνούμε με το Συμβούλιο σε σχέση με τις αποφάσεις του για τους ε, πρόσφυγες και μετανάστες. Εμείς θέλουμε αύξηση των πόρων έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, χειριστούμε το θέμα με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Αυτά λοιπόν, τα λίγα από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καρδία και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες οι υπόλοιπες ομάδες, τους συναδέλφους. Ε, μας διευκόλυνε η συμβαστική του στάση για να βρούμε λύσεις. Διαπραγματευθήκαμε συγκεκριμένα ποσά και γι' αυτό το λόγο για να υλοποιηθούν και να δαπανηθούν αυτά τα ποσά χρειαζόμαστε ισχυρά όργανα, ισχυρά θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και όλα τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, να εκτελεστεί ένας ε, προπολογισμό σωστά αν δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές και το κατάλληλο δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό τους ευχαριστώ όλους. Μία διευκρίνηση στις, στα άλλα τμήματα εκεί που μιλάμε για τη στρατηγική και τη συμφωνία στην οποία συμφωνήσαμε, δηλαδή να αντιστρέψουμε τις ε, μειώσεις που επέβαλε το Συμβούλιο, να πω το εξή. Ε, σεβαστήκαμε τη συμφωνία κύριων που έχουμε, οπότε δεν ακουμπήσαμε καθόλου την πρόταση του Συμβουλίου και ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία κυρίων gentlemen's Agreement θα τηρηθεί μέχρι το τέλο και ελπίζω κάποια στιγμή να αλλάξουμε και αυτό τον όρο Gentleman's Agreement, γιατί δεν πρόκειται μόνο για κυρίου ε, και οι κυρίε έχουν εξίσου ισχυρό λόγο. Thank you. Thank you. So, uh, we start to... Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία και αυτό είναι κάτι καινούριο για μένα, οπότε θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα ξεκινήσουμε με το 1α και το 1β, 2, 3, 4, 5 και τις ε, δαπάνες. Μετά θα προχωρήσουμε στα ειδικά μέσα, PPPS, πληρωμές, το τμήμα 1 και τα υπόλοιπα τμήματα. Κάπως έτσι θα γίνει η ψηφοφορία. Ωραία λοιπόν. Αφού έγινε η αρχή, Περνάμε στο 1α. Συμβιβαστική τροπολογία 1α. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά. Reserves. Έκον 61-38, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκόν 6139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά. Δημιουργία γραμμών. Γκουε 8243. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γκουε 8245. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Γκουε 8159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γκουε 8133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σχόλια. Γκουε 8108 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμπλ 56-64, υπέρ, κατά, αποχές, ΕΝΒΙ Ένβη 54-42, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Renew 7439 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Renew 7437 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος με νομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Renew 7437. 37 Πέρας ψηφοφορίας. 19 ψήφοι υπέρ, 18 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται δηλαδή. Μάλιστα. Είδατε. Renew 7438, 38 Υπέρ. Κατά. Νομίζω πως χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. Μάλιστα. Απορρίπτεται. EPP 7035. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γκουε 8124. Ταυτόσημη με την Badge ε, 4463. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. EPP 7033. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πράσινη 7684 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Renew 7440 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος. Με συγχωρείτε. Περνάμε τώρα στο 1β. H1β και ψηφίζουμε για το, τη συμβαστική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δημιουργία γραμμών τροπολογία GUE 8160. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στα σχόλια. Γκουε 8105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπάτζ 4086. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέρας ψηφοφορίας για το H1β, περνάμε στο H2. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία γραμμών, τροπολογία GUE 8247. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γκουε 8248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μπάτζ 4277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σχόλια. 82 8241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γκουε 80-88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενβι 54 54-64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπατζ 4486. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Badge 4412. 12 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Renew 7443. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Renew 7441. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Renew 7442. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελειώνει η ψηφοφορία για το τμήμα 2, τμήμα 3. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δημιουργία γραμμών. Γκουε 80-81. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5892, Υπέρ. Κατά. Νομίζω πως χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πράσινη 7, 6, 8, 5. Υπέρ. Μάλλον το ίδιο θα γίνει και εδώ. Εβδομήντα Α, δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε αυτή. Okay, I repeat. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. 76-85. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην Γκουε 8240. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΦΕΜ 6208. Όπως και πράσινη 7680 και ΛΥΜΠΕ 5839. Υπέρ. Κατά. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Λίμπε 5842, ταυτόσιμη με την 6218 και την 7681. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρασε. Απορρίπτεται. ΦΕΜ 6219. Ταυτόσημη με την 7682. Υπέρ. Κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Διαχωρισμός γραμμών. Λίμπε 58-90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. S&D 7393 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Λίμπε 5891 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται S&D 7392 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία για την γραμμή 3 και περνάμε στην 4. Προσπαθείτε να με αποσταθεροποιήσετε. Περνάμε στον τομέα 4, συμβαστική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πιστώσεις. Γκουε 82-39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πράσινη 76-61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αφετ 53-88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. S&D 72-48. με την badge 43-47. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. EPP 7123 με προφορική τροπολογία του εισηγητή σας έχει διανομηθεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται δημιουργία γραμμών ΦΕΜ 6211 και πράσινη 7683 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΕΚΟΝ 6120 υπέρ κατά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας Ψηφίσατε. Απορρίπτεται. Αφετ 5382. Υπέρ. Αφετ 5382. Ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αφετ 5320 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ντεβε «ΝΤΕΒΕ Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. «ΑΦΕΤ5322» και Ντεβε 5721 Α, όχι, με συγχωρείτε, λέει πρόεδρος. Ψηφίζουμε μόνο την ΑΦΕΤ 5322. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 5721. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΑΦΕΤ 5323. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άφετ 5324. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άφετ 5388. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άφετ 5390. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρινιού 7427. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για τον τομέα 4. Heading 5. Compromise. Τίτλος 5. Ποιος είναι υπέρ για το συμβιβασμό. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Δημιουργία γραμμών. Στον τίτλο 5. 42-77 από την Μπάτζη. Κατά. Αποχές. Renew. Τις παρατηρήσεις. 74-32. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αφετ 53-19. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ειδικά όργανα. Ειδικά εργαλεία. Γκουε. 81-90 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πιλωτικά προγράμματα και δράσεις, προπαρασκευαστικές δράσεις ψηφίζουμε για το πακέτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Διαγραφή γραμμών. Γκουε 8004, όπως ID 7703. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Διαγραφή γραμμών, έτσι. Γκουε 8067. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πληρωμές. Συμβιβαστική πρόταση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελειώσαμε το τμήμα 3. Περνάμε στο τμήμα 1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ψηφίζουμε το συμβασμό, συμβαστική πρόταση. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. χωριστες φιοφορίες. Ίμκο 6359. Ίμκο 6359 και ταυτοχρονα 6360. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Περνάμε στην budget, budget. Αν θέλετε να το επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε την IMCO 6359 και την 6300. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Άρχεται η ψηφοφορία. IMCO 6359, IMCO 6360. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 43-31 με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 63-59 υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. Άλλα τμήματα. Πρώτον, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε μπλοκ όλες τις τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό υπέρ, κατά, Εποχές, Εγκρίνεται. Το ελεκτικό συνέδριο. Ψηφίζουμε το συμβασμό υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Ψηφίζουμε το συμβασμό υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Επιτροπή των Περιφερειών. Συμβασμό. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ευρωπαϊκός Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Ψηφίζουν το συμβασμό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ευρωπαϊκός ε, Επιτηρητής ε, Προστασίας Δεδομένων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ψηφίζουν το συμβασμό υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. Έχουμε χωριστή ψηφοφορία τώρα για την ΑΦΕΤ 5392. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε και το κεφάλαιο αυτό και συνολικά την ψηφοφορία μας. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στις κύριες Χολμάγερ και Γκάρδια Θαβάλ. Πριν το σκάσετε, δύο λεπτάκια. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ουρέλ της Κομισιόν. Έχετε σχόλια να κάνετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αποφύγω να κάνω λεπτομερή σχόλια. Ήταν πετυχημένη η ψηφοφορία αυτή. Συγχαρητήρια λοιπόν και από τη δική μας πλευρά, ιδιαίτερα για τις δύο συγγήτριες, συνεισυγήτριες. Ποτέ, νομίζω, δεν έχω δει ψηφοφορία αυτού του θέματος να τελειώνει τόσο γρήγορα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια. Κάποιες προκαταρκτικές μόνο παρατηρήσεις. Όπως γνωρίζετε, όπως κάθε χρόνο, η Κομισιόν θα στείλει τα λεπτομερή της σχόλια για τη θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στο, στην επιστολή εκτελεσιμότητας. Αυτό θα γίνει αμέσως μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, δηλαδή τέλος Οκτωβρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη αυτή της Επιτροπής ε, που υιοθέτησαν πολλές τροπολογίες ε, στην, στις συμβαστικές προτάσεις ε, επανερχόμενοι στις αρχικές προτάσεις δηλαδή της Κομισιόν και ακυρώνοντας μειώσεις που είχαν γίνει. Επίσης χαίρομαι που οι συγκήτριες έλαβαν ε, υπόψη τις ε, αρχικές ε, παρατηρήσεις της Κομισιόν για τα προκαταρκτικά σχέδια και τα πιλωτικά προγράμματα. Και αυτό θα μας διευκολύνει στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τελευταία παρατήρηση, το προφανές λέω βέβαια, είναι πολύ φιλόδοξο το πακέτο αυτό. Εξαιρετικά φιλόδοξο θα έλεγα. Όπως και το Κοινοβούλιο, έτσι και η Κομισιόν πιστεύει ότι οι περικοπές του Συμβουλίου ήταν υπερβολικές. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαδικασία ε, συμβασμού ε, και η Κομισιόν θα παίξει επικοδομητικά το ρόλο της. Οι συγγήτριες θα ήθελαν το λόγο. Κυρία Χολμάιερ, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλή συνεργασία που είχαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας βοήθησε πάρα πολύ, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που είχαμε σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης, με τη δυνατότητα να υποβάλουμε αιτήματα. Ήταν πολύ θετικά προσκύμενοι απέναντί μας. Ε, για ορισμένε περιπτώσει, πούμε, μα είπε ότι δεν γίνεται αυτά τα κονδύλια να απορροφηθούν. Ήταν πολύ ξεκάθαρη. Θα ήθελα λοιπόν να την ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία και να πω ότι ε, σε τελική ανάλυση πρόκειται για δικά τους κονδύλια, γι' αυτό τους εύχομαι καλή τύχη το Νοέμβριο. Ναι, ναι, έγνεψε καταφατικά ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρωτού λοιπόν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, να σας υπενθυμίσω τις ακόλουθες εκδηλώσεις. Ψηφίζουμε το ψήφισμα και τις ε, τροπολογίες επί του προϋπολογισμού στις 14 Οκτωβρίου. Οι τριμερείς διάλογοι έχουν προγραμματιστεί για τις 16 ε, και 17 Νοεμβρίου. Ε, τον Οκτώβριο του στις 23 Οκτωβρίου θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια και η πρώτη ε, συνδιαλλαγή ε, είναι προγραμματισμένη για τις 4 Νοεμβρίου το απόγευμα. Επόμενη συνεδρίαση. Ναι, ναι, ναι. 7 Νοεμβρίου θα γίνει ο τριμερής διάλογος. 7 Νοεμβρίου και 16 Οκτωβρίου. Συνδιαλλαγή 4 Νοεμβρίου, όπως είπαμε. Συνάντηση συνδιαλλαγής. Ναι, η πρώτη λοιπόν συνάντηση συνδιαλλαγή 4 Νοεμβρίου το απόγευμα. Επόμενες συνεδριάσεις ε, αφορούν φυσικά τι ακροάσεις επιτρόπων. Έχουμε τον ε, κύριο Χάν την Πέμπτη, αύριο την κυρία Φερέρα και τον κύριο Τζεντιλόνι την Πέμπτη. Την επόμενη Τρίτη θα γίνει ακρόαση του κυρίου Ντομπρόφσκη. Σας ευχαριστώ πολύ.